καλοχαιρετίζω θερμά κυρίε και κύριοι. Περνάμε στο πρώτο σημείο τη ημερησία διάταξή μα. Είναι η έκθεση Μπέρμαν αυτό. Αποκάλυψη στοιχείων ε, μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένε μεγάλε εταιρείε και ομίλου. Φαίνεται σημαντικό αυτό το θέμα. Ο συνάδελφο Χάουιτ εκπροσωπεί τον συνάδελφο Μπέρμαν. Περνάμε άμεσα στην ψήφιση των προτάσεων. Έχουμε την τροπολογία 2 με προφορικέ τροποποίησεις. Ναι, εσείς τι λέτε. Συγγνώμη, είναι τώρα σε σχέση με την ε, Αντιεπιτροπή. Κύριο ε, Μπέρμαν όμω ε, δεν θα ήθελε τι προφορικέ τροποποίησει σε τμήματα. Ζήτω συγγνώμη, αλλά πρέπει να εκφραστούμε εναντίον. Ευχαριστώ. Sind vier Leute. Πρόεδρος, τέσσερις από τα μέλη. Χρειάζεστε τέσσερις κατά προφορικών τροποποιήσεων. Υπάρχουν αυτοί οι τέσσερις. Συναθρίζονται. This is every how they define solidarity. Das in the oral amendments go? Amendment one and three. Yeah. Και αυτές τις προφορικές τροποποίησεις ένα και τρία. Θα ψηφίσουμε λοιπόν. Πρώτο τμήμα λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε. Μάλιστα. Ποιοι είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Απορρίφθηκε. Σαφές. Ποιοι είναι υπέρ του δεύτερου τμήματος. Κατά απόχε, εγκρίθηκε το δεύτερο τμήμα. Για το πρώτο τμήμα λέτε εσείς. Για το δεύτερο. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν. Πάλι ξανά. Υπέρ του δεύτερου τμήματος. Είχατε υπερψηφίσει. You voted with yes. Είχατε υπερψηφίσει. That's the point. The Christian Democrats are confused and the Socialists do what they are told. Υπάρχει κάποια σύγχυση από τους μεν, οι σοσιαλιστές κάνουν ό,τι τους λένε. The Christian Democrats are method where we are is chaos, but we cannot be everywhere. Abstimmung ist geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας. 12-14 εναντίον απορρίφθηκε υπέρ του τρίτου τμήματο. Κατά αποχέ. εγκρίθηκε. Να ελέγξουμε, ωραία ελέγχουμε, άρχεται η ψηφοφορία επί του τρίτου τμήματο. Πέρας ψηφοφορία. απορρίφθηκε, το είχα πει, εν πάση περιπτώσει. And Ah, <laughs> okay. so it's uh, won by 17 to 60. 17-16 λοιπόν το αποτέλεσμα. Εγκρίθηκε. Η τροπολογία 16, ναι. Ποιοι είναι υπέρ του πρώτου τμήματος τώρα. Υπέρ του δευτέρου, όχι, λάθος, κατά του πρώτου τμήματος αποχές εγκρίθηκε υπέρ του δευτέρου τμήματος κατά αποχές απορρίφθηκε το δεύτερο τμήμα τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβιβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 24. Έχουμε και προφορική τροποποίηση εδώ. Εντάξει, λοιπόν, ωραία. Πρώτο τμήμα. Είναι σε δύο τμήματα αυτή η τροπολογία, έτσι. Έχουμε δύο τμήματα. Okay. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε με την προφορική τροποποίηση. Εντάξει, υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 26 και 27 υπέρ αυτών. Είναι ένα καλό μείγμα αυτές οι δύο. Υπέρ αυτών των δύο. Κατά αποχές εγκρίθηκαν. 28 υπέρ κατά Απορρίφθηκε. 29. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε το δεύτερο τμήμα. 30 υπέρ. Πρώτο τμήμα της 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε 31 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 36 υπέρ κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 37 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Υπέρ του δευτέρου τμήματος, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 1, υπέρ. Εντάξει, ωραία. Δεύτερο τμήμα. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 37 δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 14 υπέρ 19 εναντίον απορρίφθηκε. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Όχι, εγκρίθηκε, διορθώνει ο πρόεδρος. Εγκρίθηκε έτσι, ωραία. Εγκρίθηκε. mit 14 14 υπέρ 18 εναντίον. Πώ γίνεται αυτό, οι φιλελεύθεροι υπερψήφισαν. Τι αποτέλεσμα είναι αυτό. Ένα ε, είναι ε, Οι φιλελεύθεροι είναι αυτοί, έτσι. Τι έγινε εδώ. Τροπολογία 4 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 4 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 18 υπέρ 16 εναντίον εγκρίθηκε. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 7 υπέρ. Να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 6 και άρχεται ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορία. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ, λέει ο πρόεδρο. Θα τα ψηφίζουμε όλα ηλεκτρονικά μέχρι τέλου. εντάξει, ωραία. Ποια ήταν αυτή η 6, έτσι, ωραία. Η 7 τώρα, υπέρ, κατά, Yeah, well, you voted. Uh... Check. Να ελέγξουμε λοιπόν. Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε την 7 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Τι βλέπουμε εδώ. Μάλιστα. Καταψηφίστηκε. Αντραχ 9 dafür. 9, τροπολογία 9 υπέρ. 8 διορθώνει ο πρόεδρος, υπέρ της 8, υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 10 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. 11 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. Εγκρίθηκε διορθώνει ο πρόεδρος. Εγκρίθηκε λοιπόν. Απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε. Δεύτερη διόρθωση. 11. Έτσι. Ωραία. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. 17 υπέρ 16 εναντίον. Εγκρίθηκε κύριε. 12 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ψηφίζουμε την 12. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 17 υπέρ 18 εναντίον. Απορρίφθηκε. Έχω την εντύπωση ότι για αύξηση κάποιων μισθών κάποιοι ψηφίζουν κρυφά και μυστικά και υπερψηφίζουν. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτό το αποτέλεσμα. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 14 και 15 ομού υπέρ αυτών. Κατά αποχές εγκρίθηκαν. Υπέρ του συνόλου της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Nein, ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Μάλιστα, εγκρίθηκε η έκθεση 25 ψήφοι υπέρ 10 εναντίον. Θερμά συγχαρητήρια προς τον κύριο Μπέρμαν. Μέσω του κυρίου Χάουιτ θα κεράσει μπύρα που έδωσε σωστή ικανοποιητική επιτυχή μάχη για αυτό το θέμα. 25-10 επαναλαμβάνει ο πρόεδρος το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 25-10. Καμία αποχή. Εντάξει. Ωραία. Äh, Περνάμε τώρα στην έκθεση για την Ισλανδία. Έκθεση προόδου αναφέρεται. Και πραγματικά δημονώ να ακούσω ποιες προόδους θα μας αναφέρει ο κύριος συνάδελφος Πρέντα. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Mulțumesc, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ καλά. Και πάλι κάνουμε λόγο εδώ για την Ισλανδία, για άλλη μια φορά. Είχαμε συζητήσει για την Ισλανδία πριν από τέσσερις μήνες. Τώρα, στο μεσοδιάστημα τι συνέβη. Ήταν πολύ χρήσιμο το ότι είχαμε αυτό το διάλειμμα, το ενδιάμεσο διάλειμμα τεσσάρων μηνών. Είχαμε μια ευκαιρία να αξιολογήσουμε τις μεταβολές, τις αλλαγές ε, που επήλθαν <clears throat> όσον αφορά τις ε, εκλογές. Όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζετε, η Ισλανδία εξακολουθεί να είναι υποψήφια χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση η κυβέρνηση για την, ε, το πάγωμα, την, ας το πω έτσι, την αναβολή των διαπραγματεύσεων ε, για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει η κυβέρνηση τώρα μια μελέτη που θα συνταχθεί από το Ίδρυμα το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Μελετών στο Reykjavik. Στόχος αυτής της μελέτης θα είναι να αξιολογήσει το στάδιο στο οποίο βρίσκονται και την φάση αυτών των διαπραγματεύσεων όταν σταμάτησαν και δεν προχώρησαν πλέον. Και επίσης ε, στόχος είναι να αξιολογηθούν οι εξελίξεις στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή αυτή που έγινε, διότι οι πολιτικοί δεν επιθυμούν να λαμβάνουν κάποιες αποφάσεις προτού έχουν στη διάθεσή τους αξιόπιστα στοιχεία Προτού ακούσουν δηλαδή με άλλα λόγια τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των επαϊόντων του Ιδρύματος Ευρωπαϊκών Μελετών στο Ρέικιαβικ. Αρχικά πρώτα σε μια πρώτη φάση είχαμε κάποιες ε, διαβουλεύσεις και συζητήσεις μετά τη μελέτη του φθινοπόρου. Είχαμε την έκθεση του Πανεπιστημίου του Reykjavik, έχουμε αυτή την έκθεση που θα δημοσιευτεί τον Ιανουάριο. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι κάποιες εβδομάδες, ίσως και μήνες θα πρέπει να αναμείνουμε περαιτέρω, μέχρι ότου θα υπάρξει μια σαφής θέση και τοποθέτηση από την Ισλανδική κυβέρνηση. Με βάση ακριβώς βέβαια αυτή την έκθεση που προανέφερα. Τώρα, δεδομένων όλων αυτών, των αβεβαιοτήτων που απορρέω υπάρχει και η κοινή γνώμη. Οι πολίτες βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση του αριθμού των πολιτών που είναι υπέρ τώρα της προσχώρησης, της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 41,7% σύμφωνα με μια τελευταία σφιγμομέτρηση. Βλέπουμε 8% συνολικά αύξηση του αριθμού εκείνων που επιθυμούν πράγματι να ενταχθεί, να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ισλανδία. Ωστόσο υπάρχει ακόμα πλειοψηφία υπέρ του να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Και αυτό είναι ακριβώς το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ πολιτικά. Διότι η κυβέρνηση αποφάσισε να σταματήσουν, να παγώσουν οι διαπραγματεύσεις και να ληφθεί υπόψη πρώτα η μελέτη αυτή. Αλλά οι πολίτες όχι μόνο θέλουν να συνεχιστούν αυτές οι διαπραγματεύσεις, οι διαβουλεύσεις, αλλά όλο και περισσότερο κίνεται υπέρα της προσχώρησης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια διστακτική κυβέρνηση και έχουμε μια, ένα πληθυσμό πολίτες που ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο να προχωρήσει η ένταξη. Ενδιαφέρουσα αυτή η διαφορά. Από τότε που είχαμε την τελευταία συζήτηση υπέβαλε έκθεση πρόοδου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, όσον αφορά το 2012 ε, ε, για την Ισλανδία μέσα στο 2013. Είναι παράδοξο αυτό, διότι ο τίτλος της έκθεσης ακριβώς αφορά πρόοδο, έτσι. Την πρόοδο που επετεύχθη το 2012 για την Ισλανδία και μετά τις εκλογές στην Ισλανδία, μετεκλογικές προοπτικές. Μετά την ε, έγκριση προηγούμενης έκθεσης όπως θα θυμόσαστε που είχε αναβληθεί αρκετές φορές το θέμα αυτό δεν είχαμε ε, ε, μια τοποθέτηση. Είχαμε ψήφιση στην Επιτροπή αλλά όχι στην Ολομέλεια για αυτό το θέμα από πλευράς Ευρωκοινοβουλίου. Έχουμε λοιπόν μια έκθεση για το 2013, κάνουμε όμως λόγο για μια έκθεση πρώτου για το 2012 και το τι έχει συμβεί με το πάγωμα των εξελίξεων μετά τις ε, εκλογές, τις μετεκλογικές προοπτικές γενικά. Ο Επίτροπος Φιούλε μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να προχωρήσει στην εκκίνηση νέων διαπραγματεύσεων ώστε να επιτευχθεί μια θετική έκβαση και χαιρετίστηκε αυτή η θέση διότι είναι μια ορθολογική και επικοδομητική θέση. Από την άλλη πλευρά όμως σημειώνουμε διαφοροποιήσεις ε, και αντιδράσεις από πλευράς ε, ε, Ισλανδών που κάποιοι υπουργοί ασκούν επικρίσεις για τις τοποθετήσεις που δημοσιοποιήθηκαν. Εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι αντιδράσεις δεν είναι οι σωστότερες Σεβόμαστε τη θέση λοιπόν του Ισλανδού Πρωθυπουργού. Μια και η ίδια η κυβέρνηση και το Ισλανδικό Κοινοβούλιο δεν έχουν εγκρίνει ακόμα μια σαφή τοποθέτηση, αναμφίσιμη θέση, δεν θα πίστευα ότι θα μπορούσαμε εμείς ε, τούτων αυτών δεδομένων να αναμένουμε κάτι άλλο. Να υπάρχουν και επικρίσεις, ε, να γίνονται κατηγορίες ε, και να λέγεται δεν υπάρχει λέει σαφής θέση ε, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κτλ. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την προσοχή με την οποία έλαβαν υπόψη τις συμβουλές μου. Μία συμβαστική τροπολογία μόνο υπέβαλε, υπέβαλα που διανεμήθηκε στους κοιόδης εισηγητές. Πιστεύω δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτήν. Είναι μια συμβιβαστική τροπολογία που σε αυτήν συγκλίνουν όλες οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των συναδέφων για την επικαιροποίηση των θεμάτων για τη συζήτηση για την προσχώρηση της Ισλανδίας μεταγενέστερα στην Ένωση και επίσης φυσικά και το χρονοδιάγραμμα επιπλέον χρονοδιάγραμμα για την διαμόρφωση και εξέλιξη αυτών των διαβουλεύσεων. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά και με κάθε προθυμία και ετοιμότητα είμαι στη διάθεσή σας. Ο συνάδελφος Der Kollege da. I'm Συνάδελφος Ρούτσεκ. Μιλάω εξ ονόματος του συναδέλφου που δεν μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω, και αυτό θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κύριο Πρέντα για την πολύ ισορροπημένο ψήφισμα και για τι τροπολογίε, για την δουλειά με τι τροπολογίε, Ο κύριο Πρέντα βρέθηκε σε πολύ ιδιαίτερε συνθήκε και αναγκάστηκε να δουλέψει σε δύσκολε συνθήκε και εκτιμούμε πολύ το έργο του. Άρα, μια χώρα η οποία ε, βάζει υποψηφιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά διαλύει την ομάδα για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ασυνήθιστη κατάσταση για όλους μας. Άρα είναι σημαντικό ό,τι και να πιστεύουμε σε ό,τι αφορά τις δράσεις της ε, συντηρητικής κυβέρνησης ε, της Ισλανδίας, να δείξουμε στάση προσεκτική και να παραμείνουν ε, οι συζητήσεις ανοιχτές να μην προκαλέσουμε αρνητικές ε, αντιδράσεις, ε, σπρώχνοντας, επιβάλλοντας την συνέχιση των ε, συνομιλιών και γι' αυτό ενδεχομένως να κλείσει την πόρτα αυτή. Σε ό,τι αφορά το δημοψήφισμα, η κυβέρνηση της Ισλανδίας έχει καταδείξει ότι δεν ενδιαφέρεται για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μιας και έχει η υποχρέωση για διεξαγωγή δημοψηφίσματος, τελικά οι Ισλανδοί θα είναι αυτοί που θα αποφασίσουν τι θα κάνουν και κατά πόσον θα εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους. Και αν ε, η κυβέρνηση θεωρήσει ότι η υποβολή υποψηφιότητα μπορεί να γίνει χωρίς δημοψήφισμα, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε στους Ισλανδούς το απαραίτητο χρόνο για να διευκρινίσουν την κατάσταση. Να πω ότι πάντα υπάρχει κίνδυνος το δημοψήφισμα να είναι ένα ναι ή ένα όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τόσο ένα ναι ή όχι για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Άρα είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να είμαστε σε στενή επαφή με τους Ισλανδούς και να διεξαγάγουμε ανοιχτό διάλογο. Το θέμα της ε, ένταξης της Ισλανδίας είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση ελπίζοντας να διατηρηθεί αυτή η διακοινοβουλευτική εντολή της ε, Μικτής Επιτροπής και δεν έχουμε κύριε Βόρψε προβλήματα σε ό,τι αφορά την επικρόστατη τροπολογία. Φανμπάλεν. Κύριος Φανμπάλεν. Εκ μέρους της Άλτε, Η θέση μας μοιάζει με την του προελήσαντος. Η Ισλανδία είναι δημοκρατία, είναι καλοδεχούμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Όμω, ε, εν τέλει η κυβέρνηση και ο λαό τη Ισλανδία, θα κρίνουν πώς θα προχωρήσουν από εδώ και πέρα. Α μην του πιέσουμε. Αυτοί θα αποφασίσουν πώς θα προχωρήσουν, όπω είπα, πώς θα οργανωθούν. Η χώρα παραμένει καλοδεχούμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε το αποφασίσει να προσχωρήσει. Καλό όλους στην αίθουσα αυτή και που ενδιαφέρονται για την Ισλανδία να δουν τι μπορούμε να κάνουμε. Συναρτήσει βεβαίω και αυτόν που προτίθεται να κάνουν η Ισλανδία Ευχαριστώ κύριε Φανπάλαν. Ο Σερ Ρόπερτ. Ο πρόεδρος έφυγε. Πολύ ωραία. Λέμε στην Αγγλία ότι ε, φασούλι το φασούλι γεμίζει σακούλι ή ε, κάτι παρόμοιο και ε, θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο ο οποίο ήταν επικεφαλής της ομάδας που ασχολήθηκε με το φάκελο αυτόν. Μετά την επίσημη επίσκεψη καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν ξέρουμε τελικώς τι θέλουν οι Ισλανδοί. Και δεν ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Κατά την όψη ε, μου δεν νομίζω ότι θα αποφασίσουν να προσχωρήσουν. Κάποιοι διαφωνούν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι θέμα των Ισλανδών. δημοκρατία υπάρχει στη χώρα εδώ και πολλές δεκαετίες, από τα 50, οπότε θα ψηφίσουν και θα δούμε. Αυτό που ο εισηγητής είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι ε, στα, στις το ναι, το υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αρχίζει να είναι πιο ισχυρό. Πες συγχαρητήρια στον ε, εισηγητή, ο οποίος ήταν μερόληπτος έναντι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ισλανδών βεβαίω. Η ομάδα μου ECR θα περιμένει βλέποντας και κάνοντας Εν πάση περιπτώσει η απόφαση επαναλαμβάνω των Ισλανδών. Η ομάδα μου και εγώ είμαστε ικανοποιημένοι με τον χειρισμό του εισηγητή και τον χειρισμό των συμβαστικών τροπολογιών. Πρόεδρος, ο κ. Λάγκη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρε, ευχαριστώ εσάς και τον εισηγητή για την έκθεσή του. Να σας ενημερώσω εντάχει για δύο ζητήματα τα οποία δεν συζητήσαμε ακόμη. Το πρώτο αφορά τη μελέτη που ανέθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών όσον αφορά την κατάσταση των ενταξιακών διπραγματεύσεων και να σας πω και τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση τις πληροφορίες μας, η μελέτη θα συνταχθεί από το Ινστιτούτο Οικονομικών Μελετών του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας και γνωρίζουμε ότι θα είναι μια απλή καταγραφή των γεγονότων και δεν θα προβαίνει σε συστάσεις. Θα είναι έτοιμη αρχές του 2014 και θα συζητηθεί εν συνεχεία στο Ισλανδικό Κοινοβούλιο. Πέραν όμως αυτής της μελέτης, η Ισλανδική Συνομοσπονδία Εργασία, η Συνομοσπονδία Εμπορίου και η Ομοσπονδία των Εργοδοτών ανέτσαν και αυτές σχετικές μελέτες όσον αφορά την ένταξη που θα συνταχθεί από το Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων θα είναι έτοιμη και αυτή η έκθεση την άνοιξη του 2014. Οι τέσσερις αυτοί φορείς είναι εν γέννη υπέρ της συνέχισης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και η αντίληψή μας είναι ότι αυτό θα λέει λίγο πολύ και η σχετική έκθεση. Προσβλέπουμε λοιπόν στις σχετικέ συζητήσει με βάση αυτέ τις δύο εκθέσει, στην Άνοιξη του 2014. ενημερώσω επίση και για τις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η πλειοψηφία των Ισλανδών, 67% είναι υπέρ της διεξαγωγή δημοψηφίσματος και της συνέχισης των ενταξιακών διπραγματεύσεων. Το δεύτερο ποσοστό είναι 52%. Οι δημοσκοπήσεις πάντως δείχνουν επίσης ότι μόνο 41% των Ισλανδών είναι εν τέλει υπέρ της ένταξης. Ευχαριστώ κύριε Λάγκια. Κύριε Πρέντα, ε, θέλετε να πείτε κάτι. Χαίρομαι που καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια συνέντευξη σε ό,τι αφορά την Ισλανδία και ακόμη και μετά την απόφαση της κυβέρνησης να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις. Είχαμε ήδη να σχηματίσει μια ομόφωνη άποψη σε ό,τι αφορά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Και βλέπω λοιπόν ότι παραμένει αυτή η συμφωνία μεταξύ μα σε ό,τι αφορά την Ισλανδία. Κατά πάσα πιθανότητα, του επόμενου μήνε θα υπάρξουν κάποιε ε, αντιπαραθέσεις μεταξύ των ερευνών που έχουν ανατεθεί όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα ληφθεί σύντομα μια σχετική απόφαση. Νομίζω ότι τον, ε, την επόμενη άνοιξη θα ξεκινήσει η διαδικασία και η συζήτηση για το θέμα αυτό. Αυτό τι σημαίνει. Η Ισλανδία δεν πρόκειται να μπει στην ατζέντα της Επιτροπής μας συντόμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να ανακοινώσω την ημερομηνία για την ψηφοφορία 5 ε, Δεκεμβρίου την επόμενη εβδομάδα. Και έτσι μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη και να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Δυστυχώς η συνάδελφος η κυρία Γέγκλε δεν έχει φτάσει ακόμα και γι' αυτό θα πάμε κατευθείαν στο επόμενο θέμα. Έκθεση 2013 για το Μαυροβούνιο. Ο κύριος Τάνοκ. Εκτό μικροφώνου σχόλια του κ. Τάνοκ. Ε, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Έχω αφήσει την ομιλία μου στο γραφείο μου γιατί δυστυχώ μου είχαν πάει πει ότι δεν θα πάρω το λόγο εγώ τώρα. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος, να κάνουμε τότε πέντε λεπτά διάλειμμα να περιμένουμε την κυρία Γέγκλα και την ομιλία του κυρίου Τάνοκ. Mr. Tano? You, ready? So, colleagues, we can... Είστε έτοιμοι, συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με το 12, λοιπόν, της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση προόδου του 2013 για το Μαυροβούνιο. Και να δώσω το λόγο στον εισηγητή του κύριο Τάνοκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Μεγάλη μου τιμή που και πάλι σας παρουσιάζω την έκθεση προόδου για το Μαυροβούνιο που θα υποψήφια, κατέστη υποψήφια χώρα το 2012, τον Δεκέμβριο. Έχει κάνει σημαντικά βήματα λοιπόν προς την ένταξη. Επισκέφθηκα τη χώρα πριν από 10 ημέρες και παραγμένει ένα λαμπερό παράδειγμα το τι μπορεί να συμβεί και τι μπορεί να γίνει στα Βαλκάνια. Πριν από 7 χρόνια έγινε ένα αμφιλεγόμενο δημοψήφισμα σε ό,τι αφορά την απόσχεση από την Σερβία, μια χώρα η οποία έχει κυριαρχήσει επί πολλά, πολλές δεκαετίες και Πρέπει να ομολογήσω ότι αρχικά ήμουν αρκετά αντίστακτικό σε ό,τι αφορά το κατά πόσο μπορούσε να ακολουθήσει μόνο του ε, το δρόμο της ένταξή στο Μαυροβούνιο ως ε, ανεξάρτητη χώρα. Έκανα λάθος όμως. Ε, το Μαυροβούνιο έκανε πολιτικές, κοινωνικέ, οικονομικές μεταρρυθμίσεις, αλλά έχει ξεπεράσει και την Σερβία σε ό,τι αφορά την διαδικασία προσχώρησης οι συναντήσεις λοιπόν για την ε, εξέταση όλων των κεφαλαίων έχουν ολοκληρωθεί και τώρα παραμένουν τα κεφάλαια 23-24, τα πολύ σημαντικά σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού ε, συστήματος, θέματα καταπολέμησης οργανωμένου εγκλήματο, απάτης ε, και ούτω καθεξής. Αυτές λοιπόν οι διαπραγματεύσει θα ξεκινήσουν επισήμων τους επόμενους μήνες και από ό,τι φαίνεται το Μαυροβούνιο ενδεχομένω ε, να είναι το επόμενο μέλος, το επόμενη χώρα που θα προσχωρήσει στην Ένωση. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αυτό πριν από το 2021 το νωρίτερο. Είναι μικρό και πάρα πολύ όμορφο το Μαυροβούνιο στα Δυτικά Βαλκάνια. Θα πρέπει να τονίσω πόσο θετικές είναι κάποιες ενδείξεις ε, που αναφέρονται στην έκθεσή μου. Μεγάλη συνένεση καταρχάς σε ό,τι αφορά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και η πιο ε, ισχυρή, αν θέλετε, η πιο ε, μεγάλη πολέμη της κυβέρνησης είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπάρχουν και κάποια αρνητικά στοιχεία. Ελευθεροτυπία υπάρχει. Ε, ποικιλία στην κοινωνία υπάρχει. Αλλά για πρώτη φορά είδα κατά τις επισκέψεις μου ότι κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις και κάποια μέσα ενημέρωσης ε, καλύπτονται, μάλλον φιλοξενούνται σε χώρους της πρώην αντιπολίτευσης. Υπάρχουν λοιπόν πολύ λίγες ευκαιρίες σε ό,τι αφορά και την δημιουργική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Αυτό ίσως να έχει και αντίκτυπο στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Υπάρχουν ε, διάφορες ε, ε, περιπτώσεις και υποθέσεις βίας κατά των δημοσιογράφων, οι οποίες αναφέρονται και στις εφημερίδες. Υπάρχουν όμως και βασικά ζητήματα κατά πόσον έχει εξουσία ο τύπος να παραπλανήσει το κοινό. Και αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που αποσχολεί γενικότερα τους δημοσιογράφους. Άρα λοιπόν οι εσωτερικοί διχασμοί μεταξύ των Μαυροβούνιων ενδεχομένως να επιβραδύνουν την διαδικασία προσχώρησης. Παρά το γεγονό ότι η κυβέρνηση λοιπόν εφαρμόζει τι μεταρρυθμίσεις και η κοινωνία των πολιτών ασκεί επικοδομητική κριτική. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά θα πρέπει να λάβουν χώρα σε κοινοβουλευτικέ διαδικασίε, αλλά φαίνεται ότι περιορίζονται εκτός της ε, κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Η έκθεση ακολουθεί την συνηθισμένη, το συνηθισμένο σύστημα σε ό,τι αφορά την δομή τη, τα θέματα είναι λίγο πολύ τα ίδια με πέρσι και πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν σε ό,τι αφορά το εκλογικό, εκλογική νομοθεσία, σε ό,τι αφορά το δικαστικό σώμα. Υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ότι στις επερχόμενες εκλογές από τους βουλευτές του ε, κεντρικού εισαγγελέα θα επιφέρει μια σημαντική αλλαγή στο κράτος δικαίου επίσης θα πρέπει να καταπολεμηθεί αυτή η κουλτούρα της ατιμορρησίας σε ό,τι αφορά θέματα διαφθοράς και απάτη σε υψηλά επίπεδα. Κάποια μέλη του κυβερνώντος κόμματος καταχράστηκαν τα δημόσια ταμεία σε ό,τι αφορά τις προεδρικές εκλογές. Το αναφέρω αυτό. Δεν θέλω ωστόσο να επικρίνω οτιδήποτε, γιατί αυτό είναι στα χέρια του δικαστικού σώματος και το δικαστικό σώμα θα πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Δεν είναι θέμα αυτοκοινοβουλευτικής έκθεσης σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των μειονοτήτων τώρα και σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τους ΛΟΑΤ, τους Ρώμα και άλλα θέματα ισότητα των φύλων, σημειώνει, εξακολουθεί να σημειώνει πρόοδο το Μαυροβούνιο. Μόνο δύο άνδρες έχουν δηλώσει ανοιχτά στο Μαυροβούνιο από ό,τι φαίνεται και προφανώς ε, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ θα πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά. Πέρα από το εξαιρετικό έργο της αστυνομίας ε, σε ό,τι αφορά τις, ε, τα δύο gay pride που έγιναν προσφάτως. Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι οι φιλοδοξίες σε σχέση με το ΝΑΤΟ. Πιστεύω ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα ενίσχυε τις μεταρρυθμίσεις του Μαυροβούνιο και θα επιτάχυνε και τις διαπραγματεύσεις ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Υπουργός Άμυνας στο Μαυροβούνιο ε, συμβάλλει βασικά σε ό,τι αφορά την κοινή πολιτική, πολιτική και πολιτική άμυνας. Και γι' αυτό λοιπόν σκοπεύω να καταθέσω μία τροπολογία σε ό,τι αφορά την έκθεση. Άρα, συνολικά είναι καλέ οι καλά τα νέα για το Μαυροβούνιο. Καλωσορίζω τις ε, παρεμβάσει και τι τροπολογίε των ε, συναδέλφων και ελπίζω να μπορέσουμε να καταρτήσουμε και συμβιβαστικέ τροπολογίε σε ό,τι αφορά και την ψηφοφορία στα πλαίσια τη Επιτροπή μα, Ελπίζω τον Γενάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ για την παρουσίαση Τη έκθεσης προόδου για το Μαυροβούνιο να δώσω τώρα την δυνατότητα και στους σκιώδεις εισηγητές να συζητήσουν, να καλωσορίσουμε και την κυρία Γέκλε, αλλά θα συνεχίσουμε πρώτα την έκθεση για το Μαυροβούνιο, καθότι δεν μπορούμε να διακόψουμε. Από το ΕΛΚ, λοιπόν, έχουμε την κυρία Μπεσαβίτς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως πάντα, ο κύριος Στάνοκ από πλευράς του συνέταξε μια καλή έκθεση που είναι πολύ ισορροπη, ισορροπημένη. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Με παρακολουθείτε, μπορείτε να με ακούσετε. Μπορώ να μιλήσω και σλοβακικά, αν το προτιμάτε. Λοιπόν, <clears throat> συνεχίζει στα σουηδικά η κυρία Ιβρισάβιτς. Θέλω να ευχαριστήσω όπως είπα τον κύριο Τάνοκ για μια καλή ισορροπημένη έκθεση. Το ένα ή άλλο σημείο θα ήθελα να εξετάσουμε επιμέρους. πολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος είναι κύριες προτεραιότητες, αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο για το Μαυροβούνιο, ισχύει για το σύνολο των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο θα πρέπει να ενδιαφερόμαστε για αυτά τα θέματα. Υπάρχουν αιτήματα και απαιτήσει όσον αφορά τις χώρες ε, των Δυτικών Βαλκανίων μετά την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το Μαυροβούνιο κατά το παρελθόν είχε καταβάλει προσπάθειες, ήταν έντονα υπέρ. Ο κύριος Τένοκα το επισημαίνει αυτό το θέμα στην έκθεσή του. Θα ήθελα να δούμε και να μεριμνήσουμε παράλληλα να προχωρήσουμε όπως γίνεται και σε άλλες εκθέσεις για αυτά τα θέματα. Με την ίδια διατύπωση, το ίδιο μήνυμα πρέπει να σηματοδοτήσουμε και να αποστείλουμε σε όλες τις εκθέσεις μας, διότι τα εγκλήματα του οργανωμένου εγκλήματος δεν αφορούν μία και μόνο συγκεκριμένη χώρα, είναι διασυνοριακό αυτό το φαινόμενο και πλήττει και τα παιδιά που είναι θύματα. Γι' αυτό θα ήθελα λοιπόν να έχουμε την ίδια διατύπωση σε τέτοια εδάφια. Τώρα, για το θέμα των ελευθεριών του τύπου και των μέσων ενημέρωσης. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους και να εργάζονται μέσα σε ένα καθεστώς ελευθερίας. Ακούγοντας αυτά τα οποία αναφέρονται, έχω την εντύπωση ότι και οι ίδιοι δημοσιογράφοι επομίζονται συγκεκριμένες ευθύνες που ίσως όμως στα Βαλκάνια δεν γίνεται αυτό κατανοητό όπως στις δικές μας χώρες. Ελευθερία του τύπου σημαίνει στα Βαλκάνια ότι έχουν την απόλυτη ελευθερία οι δημοσιογράφοι να γράφουν οτιδήποτε επιθυμούν και να συντάσσουν και να λένε ό,τι θέλουν. Όμως πρέπει να μεριμνήσουμε να εξευρίσκονται οι σωστές διατυπώσεις με ισόρροπο τρόπο, διότι ελευθερία σημαίνει ότι ταυτόχρονα και ευθύνη και υπευθυνότητα από πλευράς τους. Από την άλλη πλευρά πρέπει να πω ότι κάποια γεγονότα, κάποια συγκεκριμένα θέματα θα ήθελα να επικαιροποιηθούν. Λέγεται στην έκθεση ότι καταβάλει περισσότερες προσπάθειες στο Μαυροβουνίο υπέρ των μειονοτήτων. Η Ρωμά, η Τσιγκάνη και η εντό εισαγωγικών Αιγύπτη Τσιγκάνη πάλι με άλλη ονομασία. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι το Μαυροβούνιο κατά το 2012 είχε ξεκινήσει και είχε συντάξει ένα πρόγραμμα δράσης για αυτές τις μειονότητες. Θα δώσω συνέχεια σε αυτό και θα μπορέσω έτσι να φωτίσω τα γεγονότα αυτά και να τα δω πιο συγκεκριμένα. Η αντιπολίτευση και την έκθεση ενδεχόμενα μπορεί να την αμφισβητήσει και μπορεί να τεθεί και κατά του κυρίου Τένοκ και να πει ότι εξοραίζονται τα πράγματα υπερβολικά. Όμως θα ήθελα να εκφραστώ υπέρ του να υποστηρίξουμε τον συνάδελφό μας αν η έκθεση αυτή είναι ισορροπημένη εναντί και εκθέσεων άλλων χωρών ή εναντί της Σερβίας για παράδειγμα, θα μπορούσε να εκφράσει την ικανοποίησή τη η αντιπολίτευση για το ότι το Μαυροβούνιο σε σχέση με άλλε χώρε ε, παρουσιάζεται υπό ένα θετικό φω. Όμω το Μαυροβούνιο δεν ισχύει αυτό. Τμήματα τη αντιπολίτευση δεν συμφωνούν ούτε και με αυτό, με το να παρουσιάζεται μια θετική εικόνα τη κυβέρνηση και τη χώρα. Παρακαλώ την έκθεση να την υποστηρίξουμε γιατί είναι πράγματι ισορροπημένη. Ευχαριστώ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 είναι πολύ ισορροπημένο το σχέδιο έκθεσης και επικεντρώνεται σε σημαντικά θέματα. Ο κύριος ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στις μεταρρυθμίσεις προς ε, κατεύθυνση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζεται και το άνοιγμα κεφαλαίων όπως ε, του 23 και του 24 στις ε, απότερες διαπραγματεύσεις. Όμως θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες σε θέματα τα οποία δεν καλύπτει ο κύριος Τάνοκ. Και αυτά τα θέματα έχουν τεράστια σπουδαιότητα. Για παράδειγμα, <clears throat> την χρηματοδότηση που πρέπει να είναι στη διάθεση να διασφαλίζεται σε μικρότερες και μη κεντροποιημένες οργανώσεις και συλλόγους των πολιτών. Θα πρέπει το Μαυροβούνιο να συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες υπέρ μιας πολιτικής ισότητας, ώστε η υποεκπροσώπηση των γυναικών για παράδειγμα στο κοινοβούλιο να αντιμετωπιστεί ή σε ηγετικέ θέσει, ή σε υπεύθυνε θέσεις για την λήψη αποφάσεων στον δημόσιο τομέα. Ίσως και ίδιος μισθός ε, είναι και αυτό σημαντικός στόχος. Φυσικά από πλευρά σοσιαλδημοκρατών είναι σημαντικό για τα θέματα των εργατικών ενώσεων και συνδικάτων θα καταθέσουμε μια αντίστοιχη τροπολογία. Όπως είπαμε, είναι μια πολύ καλή ισορροπημένη έκθεση και μπορεί να βελτιωθεί με κάποιες τέτοιες προσθήκες από πλευράς μας. Σας ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρούτσεκ. Για την ομάδα των Άλντε τώρα έχετε εσείς τον λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα <clears throat> να υποστηρίξω και να αναγνωρίσω τις προσπάθειες που κατέβαλε ο εισηγητής μας κύριος Τάνοκ για να καταφέρει να καταλήξει σε μια ισορροπημένη φιλική, επικοδομητική, με κίνητρα έκθεση, με επικοδομητικό χαρακτήρα για το Μαυροβούνιο. Ξενόματος τη της μου, εγώ προσωπικά μπορώ να πω ότι θεωρούμε ότι το Μαυροβούνιο με αργούς βέβαια ρυθμούς, όμως προχωρεί και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που έχει επομιστεί για την ε, προσχώρηση, την ένταξη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ε, γραφειοκρατίας ε, και να αντιμετωπιστεί σε πολλά επίπεδα. Έχουμε θεσπίσει μετά από μια σύντομη ε, ταραχώδη περίοδο μετά τις ε, προεδρικές εκλογές μια νέα φάση. Τώρα το Κοινοβούλιο εργάζεται με πλήρης ικανότητες και δυναμικό και υπό το πνεύμα της ε, λειτουργικής δημοκρατίας σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο. Η προσπάθεια να επιτελεστούν, να υλοποιηθούν μεταρρυθμίσεις είναι εξόφθαλμη. Σε θέματα όπως τις δημόσιες προμήθειες, τα θέματα εταιρικού δικαίου, πνευματικής ιδιοκτησίας, μέσα του τύπου και της ενημέρωσης, φορολογίας, βιομηχανικής πολιτικής, έχει επαρκώς προοδεύσει το Μαυροβούνιο και συνιστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να αρχίσουν να ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν ε, και εμείς από πλευράς όπως και ο εισηγητής προσθέτουμε τη φωνή μας υπέρ αυτού. Αναφέρθηκαν και άλλα θέματα ως αρχές που θα πρέπει να συνοδεύουν τις προσπάθειες του Μαυροβουνίου κατά το επόμενο διάστημα. Είναι σημαντικό ένα ευρύτερο πρόγραμμα δράσεων να αναλυφθεί από το Μαυροβούνιο ώστε να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις υπό ένα καθεστώς κράτους δικαίου με τις βέλτιστες προδιαγραφές για να ανοίξουν και τα κεφάλαια 23 και, 22, 23 και 24. Σε σχέση με αυτά σημαντικές μεταρρυθμίσεις και προσπάθειες όπω όπως η καταπολέμηση της ε, διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος πρέπει να τύχουν συνέχεια. Προσθέτω και εγώ τη φωνή μου στο να μπορέσουν να ανοίξουν το δυνατόν ταχύτερα νέα κεφάλαια και να δοθεί νέα προώθηση στις ε, μεταρρυθμίσεις. Είναι σημαντικό ότι η οικονομική και, κοινωνική, η οικονομική και κοινωνική κατάσταση στη χώρα χαρακτηρίζεται με ένα ποσοστό, από ένα ποσοστό ανεργίας περίπου γύρω στο 20% η κοινωνία των πολιτών έχει ενταχθεί και έχει ε, προχωρήσει σε αρκετές διεργασίες. Είναι όμως σημαντικό αυτή η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των οργανωμένων πολιτών να βελτιωθεί ακόμα περαιτέρω. Και στο περιφερειακό πλαίσιο ο ρόλος του Μαυροβουνίου θα πρέπει να αναγνωριστεί και να προαχθεί. Τέλος, ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι. Να πω <clears throat> ότι ο καθορισμός της συνοριακής γραμμής ε, και η επίλυση μεθοριακών θεμάτων συνόρων, όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση της Επιτροπής, είναι σημαντική υπόθεση. Το Μαυροβούνιο από κοινού με τους γείτονες ε, θα πρέπει να προσπαθήσει τα θέματα που εκκρεμούν όσον αφορά την χάραξη και τον καθορισμό συνόρων αμοιβαία να προχωρήσει για να αρθεί έτσι ένα μείζον εμπόδιο, να μην έχουμε προβλήματα μεταξύ των χώρων αυτής της περιοχής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τους ε, πρασίνους ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξ ονόματος Λούνατσεκ θα παρέμβω. Ε, κύριος ε, Ντεμές Μέκερ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τένοκ για αυτή την έκθεση. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα έπρεπε να αναφέρουμε βέβαια. Να επανέλθω πρώτα στην ψήφιση στην Ολομέλεια για την έκθεση του Μαυροβουνίου τον Απρίλιο μετά τις προεδρικές εκλογές. Εκφράζαμε τη θλίψη μας ε, γιατί δεν μπορούσε να επιτευχθεί υποστήριξη για την τροπολογία που είχαμε καταθέσει για τα επίμαχα θέματα αμέσως μετά τις εκλογές. αυτή μας την τροπολογία είχαμε θέσει το θέμα των μεγάλων προβλημάτων παρατυπιών ε, και ολισθημάτων που είχαν σημειωθεί για την χρήση και δημοσίων κονδυλίων σε αυτή την εκστρατεία. Θα μπορούσαμε να επηρεάσουμε τις εξελίξεις στο Μαυροβούνιο, αλλά αποτύχαμε ως Ευρωκοινοβούλιο να το πράξουμε αυτό. Τώρα το θέμα της καταχώρησης ψηφοφόρων και το θέμα της χρήσης ε, κονδυλίων των φορολογουμένων ανεβρίσκεται στην έκθεση του κυρίου Μένα, αλλά δεν υπάρχει επαρκής πίεση επ' αυτών. Μια κοινοβουλευτική επιτροπή διακριβωτική δεν ήταν σε θέση να υιοθετήσει συμπεράσματα επ' αυτών. Και λέει ΜΑΗ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η δικαστική συνέχιση αυτών των πραγμάτων απομένει να διασφαλιστεί. Δεν είναι μικρολεπτομέρειες αυτά τα θέματα, συνάδελφοι. Είναι θέματα που αφορούν τα θεσμικά όργανα του Μαυροβουνίου και τη δημοκρατία. Αυτό που αμφισβητείται είναι αν συμμορφώνεται αυτή η χώρα με θεμελιώδη πολιτικά κριτήρια. Πρέπει να είμαστε κάθετοι και απόλυτα σαφείς επ' αυτού του θέματος. Είμαστε εμείς ε, κατά του να επαναληφθούν οπωσδήποτε, να μην επαναληφθούν τέτοιου είδου συμβάντα στο μέλλον. Δεύτερο, ασφάλεια δημοσιογράφων και εκείνων που προσπαθούν να διασφαλίσουν ανεξάρτητες υπηρεσίες του τύπου. Έχουμε πληροφορίες ότι η κατάσταση δεν βελτιώνεται, αλλά επιδεινώνεται. Όλο και περισσότερες απειλές εκτοξεύονται κατά δημοσιογράφων και αναμένουμε και πάλι εδώ για την αρμόζουσα δικαστική συνέχεια, δέουσα δικαστική συνέχεια που πρέπει να δοθεί. Αυτές οι ελευθερίες είναι θεμελιώδους σημασίας για τα πολιτικά κριτήρια και τη συνέχεια που θα δοθεί. Είναι καλό το ότι υιοθέτησε την βελτίωση όρων διαβίωσης των ε, ε, ομοφιλοφίλων ε, η κυβέρνηση. Αλλά πρέπει να δούμε πέρα από τα χαρτιά τι γίνεται. Ένας από τους ενεργότερους εκπροσώπους αυτής της κοινότητας έτυχε ασύλου στον Καναδά. Πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό αν όλα πάνε καλά στο Μαυροβούνιο. Χρειάζονται λοιπόν περισσότερες προσπάθειες. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για αυτό το κείμενο. Θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες επί των θεμάτων που προαναφέρει αναφέρθηκαν και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία μαζί του. Ευχαριστώ. Google Group, Mr. Ευχαριστώ από την Google, κ. Φουλιανίτς. Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Τάνο και την ισορροπημένη και τίμια έκθεση. Τίμια ενώ ότι καλύπτει τα περισσότερα βασικά στοιχεία και ζητήματα που αφορούν το Μαυροβούνιο και τα λέω φιλική, προσπαθεί να είναι ενθαρρυντική προς τη χώρα, το οποίο πρέπει να είναι και ο ρόλος μιας καλής έκθεσης. Ο σκοπός δεν είναι να αξιολογήσουμε, να δικάσουμε τη χώρα, αλλά να τη βοηθήσουμε. Το Μαυροβούνιο είναι μια μικρή χώρα με πληθυσμό 600.000 ανθρώπων, αλλά μια αρκετά σύνθετη χώρα, πολύπλοκη θα έλεγα, λόγω της ε, σύνθεσης του πληθυσμού, των κατοίκων, των θρησκειών, αλλά και της ιστορίας. Η πολυπλοκότητα αυτή, εν τούτης, δεν είναι στη ρίζα των περισσότερων προβλημάτων της χώρας. Γιατί δεν υπάρχει εθνικισμός, ε, ούτε εθνικός, ούτε ε, θρησκευτικός φανατισμός. Από τη δεκαετία του 90 κυβερνά το ίδιο κόμμα σε μια χώρα μισού εκατομμυρίου και κάτι. Αυτό σημαίνει ότι ένας μικρός κύκλος ανθρώπων, είναι σχεδόν μια οικογένεια, κινεί τα νήματα. Κάτι το οποίο αναπόφευκτα έχει οδηγήσει σε διαφθόρα, οργανωμένο έγκλημα να έχει σχωρήσει στους κόλπους της κυβέρνησης. Παρατηρούμε επίσης τα εθνικά περιουσιακά στοιχεία να πολλούνται σε κυκλώματα ξεπλήματος ε, μαύρου χρήματος και το καθεξής. Γίνεται βέβαια προσπάθεια στο Μαυροβούνιο, κατάλληλο αυτό, αυτό είναι αλήθεια και εν ε, με τρόπο επιτυχημένο. Όμως το βασικό πρόβλημα είναι η κομματοκρατία, η οποία είναι μία από τι βασικέ ε, ασθένειε τη χώρα μετάβασης. Το Μαυροβούνιο δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Το ζήτημα αυτό θεωρώ ότι πρέπει να αναφερθεί με σαφήνεια και συνεχώς σκοπεύω να καταθέσω κάποιες τροπολογίες. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν προβλήματα τα οποία αναφέρει η έκθεση με σαφήνεια. Το Μαυροβούνιο κάποια στιγμή θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει θέματα όπως η παντελής έλλειψη βιομηχανίας στην χώρα, ό,τι υπήρχε πριν τη δεκαετία του 90 καταστράφηκε, μετά είναι η υψηλή ανεργία, είναι ζητήματα δηλαδή που η χώρα πρέπει να αντιμετωπίσει και εν των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα απολύτως με τον εισηγητή ότι τα κεφάλαια 23 και 24 πρέπει να ανοίξουν διότι είναι οι τομείς στους οποίους η χώρα έχει πετύχει τα περισσότερα αλλά και που αναμένεται να κάνει τα περισσότερα. Είμαστε υπέρ λοιπόν. Τσεκ, ευχαριστώ. Πρόεδρος μετά του κοιόδης εισηγητές. Έχω εδώ δύο πλέον ομιλητές. Κύριος Κούκαν, πρόεδρος και της αντιπροσωπείας. Πρόεδρε, συγχαρητήρια καταρχήν στον κύριο Τάνοκ για την έκθεσή του για το Μαυροβούνιο. Καλή έκθεση. Θα περιοριστώ σε λίγα σχόλια. Εν γέννη, εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι προχωρά προς τον μπρός η ενταξιακή διαδικασία. Πρέπει όμως να είμαστε ακόμη πιο απαιτητικοί για να προχωρήσουμε ακόμη πιο γρήγορα και με τρόπο ακόμη πιο ουσιαστικό. Θα ήθελα λοιπόν να παρακινήσω την κυβέρνηση τη χώρα να συνεχίσει τον ίδιο δρόμο με την ίδια ταχύτητα, ιδιαίτερα όσον αφορά την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που είναι κρίσιμη σημασία και πρέπει να πάνε σε βάθο. Κράτο δικαίου και σχετικές μεταρρυθμίσεις. Εδώ πρέπει να προχωρήσουμε με την ίδια επιμονή, γιατί τα κεφάλαια 23 και 24 είναι πολύ σημαντικά. Ο αγώνας κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος πρέπει και αυτός να συνεχιστεί. Και οι βασικές ε, υποθέσεις πρέπει κάπου να καταλήξουν. Σύμφωνα με τον κύριο Τάνοκ, όσον αφορά την απαραίτητη καθυστέρηση της έκδοσης πρωτοδίκων αποφάσεων ή υποθέσει οργανωμένου εγκλήματος. Ελευθερία έκφραση και ελευθερία τύπου και αυτές πρέπει να προστατευθούν. Θα ήθελα να θυμίσω ότι οι επιθέσει κατά δημοσιογράφων είναι απαράδεκτες και καλό τι αρμόδιες αρχές να δείξουν τον δρόμο και να προχωρήσουν σε ενδελεχεί έρευνε συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ενταξιακή διαδικασία και στις μεταρρυθμίσεις. Και αυτές είναι κρίσιμες σημασίας. Πρέπει να στείλουμε το μήνυμα με τρόπο διαφανή προς την κοινή γνώμη. Χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση και περισσότερη πληροφόρηση προς τους πολίτες της χώρας. Τέλος, εξίσου σημαντικό, τα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα πρέπει να τύχουν σοβαρή αντιμετώπιση από την κυβέρνηση. Θίγονται όλα αυτά βεβαίω στην έκθεση του κυρίου Τάνο και εγώ να προσθέσω μόνο την ανάγκη το κλίμα για τις επιχειρήσεις να βελτιωθεί και να παγιωθεί. Επίσης θα χρειαστεί μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση με περισσότερη ανοχή για τη βοσνιακή μειονότητα και τους Ρωμά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Έντουαρτ. Λόγο στον κύριο Στία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον κύριο Τάνοκ για την πολύ καλή έκθεση, η οποία καταδεικνύει με σαφήνεια την πρόοδο που έχει πετύχει το Μαυροβούνιο το τελευταίο χρόνο. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι και πιστεύω ότι το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24 θα αποτελέσει το σωστό πλαίσιο για τις περαιτέρω αποφάσει. αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα την οικονομική κατάσταση. Να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη δική της έκθεση τόνισε και αυτή ότι τα δικαιώματα APR εναρμονίζονται σε μεγάλο βαθμό με το κινητικό κεκτημένο. Και πάλι όμως θα πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις προκειμένου να εφαρμοστούν όλα αυτά καλύτερα στην πράξη. Και υπό την έννοια αυτή, σε ό,τι αφορά τα, τις εταιρείε. Ε, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα πνευματικών ε, δικαιωμάτων, της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις και θα κάνουμε κάποιες ε, τροπολογίες ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Να καλωσορίσω επίσης το άρθρο 4 που μιλά για την ε, μεγαλύτερη πολιτική βούληση που θα πρέπει να υπάρχει προκειμένου να εξηγηθούν με καλύτερο τρόπο στο λαό του Μαυροβουνίου τα στοιχεία των διαπραγματεύσεων. Και υπό την έννοια αυτή λοιπόν πιστεύω ότι αυτό θα αποτελούσε ένα ωφέλιμο βήμα. Κλείνοντας, να πω ότι το Μαυροβουνίο έχει πετύχει σημαντική πρόοδο και η πρόοδος αυτή είναι ασφαλώς θετική. Και αυτό αντικατοπτρίζεται και αποτυπώνεται καλά στην έκθεση. Ευχαριστώ, κύριος. Ευχαριστώ, κύριε Στήρ. Ο κύριος ε, Πίκουλα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω όλες τις αποχρώσεις που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση. Να συγχαρώ λοιπόν τον εισήγητη να τονίσω επίσης ότι το δημοψήφισμα του 2005 δεν ήταν αμφιλεγόμενο. Αλλά οι κανόνες αναφορικά με το δημοψήφισμα επιβλήθηκαν στους Μαυροβούνιους. 55% προσέλευση έπρεπε να υπάρχει για να ανακηρυχτεί η ανεξαρτησία. Άρα, υπήρξε αυτή η προσέλευση και ακόμα και πριν το δημοψήφισμα σε ό,τι αφορά τις ε, συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση υποστήριζαν την εξαρτησία τους. Ε, να τονίσουμε ότι είναι μεγάλη δυναμική του Μαυροβουνίου σε ό,τι αφορά την πολιτική της περιφέρειας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ θετικό το περιβάλλον στη χώρα. Πρόκειται για τη μοναδική χώρα στην περιοχή που έχει αρχίσει τέτοιες συνομιλίες και διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει όμως να συντονιστεί η δράση και με τις άλλες περιφερειακές μας δράσεις για να μην υπάρχουν επικαλύψεις. Τα κεφάλαια για την Κροατία είναι πολύ σημαντικά. Και τα κεφάλαια 23-24 είναι πολύ σημαντικά ασφαλώς για όλες τις υποψηφίες χώρες. Έχει κλείσει δύο κεφάλαια, έχει benchmarks για άλλα έξι κεφάλαια του Μαυροβούνιου. Να σας υπενθυμίσω ότι πριν από 10 χρόνια συμφωνήσαμε επί ενός προσωρινού καθεστώτος για τα σύνορα μεταξύ Κροατίας και Μαυροβουνίου. Οι εμπειρίες με την Κροατία σε ό,τι αφορά το θέμα των συνόρων είναι κάτι με το οποίο πλέον έχουμε εμπειρία. Και το Μαυροβούνιο, η γειτονική αυτή χώρα, θα πρέπει να έχει και ένα δικό χάρτη, το οποίο θα πρέπει να καταρτιστεί εγκαίρως. Και θα πρέπει λοιπόν το θέμα αυτό να έχει επιληθεί πριν την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσω και πάλι το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Λάγκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω λίγο σε ό,τι αφορά και τις δικές μας σκέψεις, σε ό,τι αφορά τα περίφημα κεφάλαια 23 και 24, σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου. Θα ξέρετε ότι τα παρουσιάσαμε στα κράτη-μέλη την προηγούμενη εβδομάδα. σε ό,τι αφορά τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για πρώτη φορά θέσαμε ενδιάμεσα benchmarks τέτοια ορόσημα Πρώτη φορά λοιπόν ακολουθούμε αυτή τη νέα προσέγγιση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτά τα ενδιάμεσα benchmarks καλύπτουν ένα πολύ ευρύ φάσμα των πτυχών του κράτους δικαίου στο Μαυροβούνιο. Επίσης, αυτά τα ενδιάμεσα ορόσημα δεν είναι νέα στοιχεία ουσιαστικά, προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από το σχέδιο δράσης, άρα δεν αποτελούν ένα καινούριο παράγοντα που προκαλεί έκπληξη στο Μαυροβούνιο. Θα ολοκληρωθούν και ελπίζουμε το κεφάλαιο να μπορέσει να ανοίξει στη διακυβερνητική συνάντηση στις 18 Δεκεμβρίου. Θα έπρεπε επίσης να διευκρινίσω στο σημείο αυτό ότι όταν καθορίσαμε αυτά τα ενδιάμεσα ορόσημα, όταν δουλεύουμε επί του σχεδίου δράσης, αναμένουμε αποτελέσματα από το Μαυροβούνιο. Δεν πρόκειται για κάτι το οποίο τίθεται τώρα για δύο χρόνια δεν συμβαίνει τίποτα και μετά πρέπει να πληρώνται όλοι οι όροι. Όχι. Θέλουμε οι όροι αυτοί να πληρούνται, οι ενέργειες αυτές να γίνουν άμεσα και θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση σε εξαμηνιαία βάση. Θα υποβάλουμε και σχετικές αναφορές προς το Συμβούλιο. Τι άλλο προτείνουμε στην, στο σχέδιο κοινή θέση. Αν η πολιτική κατάσταση στο Μαυροβούνιο τροποποιηθεί, ενδεχομένως να προτείνουμε τροποποίηση και των ενδιάμεσων αυτών benchmarks και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Συνολικά λοιπόν στην ε, παρουσίασή μας και στην επικοινωνία μας με το Μαυροβούνιο επαναλαμβάνουμε αυτό που είπατε και εσείς εδώ, ότι ασφαλώς χρειάζεται υψηλή πολιτική βούληση για να, να επιτευχθούν όλα αυτά. Χωρίς την πολιτική βούληση δεν πρόκειται να ολοκληρώσουν αυτές τις διαδικασίες τις οποίες και προβλέπουμε. Ανοίγοντας όμως τα κεφάλαια αυτά, αυτό ενδεχομένως είπα να γίνει στις 18 Δεκεμβρίου, μπορεί να δοθεί η δυνατότητα να ανοίξουν και άλλα κεφάλαια. Τα κεφάλαια 23-24 είναι καθοριστικά για την συνέχιση της ε, διαδικασίας των διαπραγματεύσεων. Αν ανοίξουν αυτά τα δύο κεφάλαια, θα ε, επιτρέψει αυτό στο Μαυροβούνιο να συνεχίσει και με τα άλλα κεφάλαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε, κύριε Λάγκε. Να δώσουμε επειδή πρέπει να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Γέγκλε, να δώσω το λόγο στον κύριο Τάνοκ να κάνει κάποια σύντομα καταλητικά σχόλια. Σε ευχαριστώ πρόεδρε. Φυσικά είχαμε και προτάσεις από πραγματικά πραγματογνώμονες ε, από την περιοχή αυτή. Και καλό χαιρετίζω επίσης ε, τις παρατηρήσεις ε, της συναδέλφου Ιζιτ Συμφωνώ να χρησιμοποιούμε την ίδια παρόμοια διατύπωση σε όλες τις εκθέσεις για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τις υποψήφιες χώρες. Να ακούγεται το Κοινοβούλιο χρησιμοποιώντας μία ενιαία φωνή και τοποθέτηση αν θέλετε να υπάρξει λοιπόν μια τροπολογία να κατατεθεί για τον εναρμονισμό της ορολογίας της διατύπωσης, συμφωνώ. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το α, Μαυροβούνιο όσον αφορά την ανεύθυνη δημοσιογραφία και την ε, επικίνδυνη δημοσιογραφία. Φυσικά πρέπει η ασφάλεια των δημοσιογράφων να διασφαλίζεται από τις δυνάμεις του νόμου. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχουν δικαίωμα τιμωρησίας να επιτίθενται κατά ιουδήποτε, ακόμα και κατά ευρωβουλευτών. Ο ίδιος εγώ υπέστη σε επιθέσεις ε, και ε, ακούστηκαν τέτοιες επικρίσεις ε, και σε σχέση λέει και με πληρωμές από πλευρά της ίδιας της κυβέρνησης. Θα έπρεπε τέτοιου είδους τοποθετήσεις και ισχυρισμοί να καθοδηγούν ενώ καταλήγουν στα δικαστήρια. Ε, ίσως επειδή είμαι συντηρητικό έγιναν αυτά, όμως εν πάση περιπτώσει καλωσορίζω την σκέψη του προγραμματος δράσης για τους ε, Αθηγάνους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να γίνει κάτι για τους Ρωμά τους Τσιγκάνους. Και για τα σχόλια άλλων συναδέλφων από πλευρά Ροτσεκ έγιναν σχόλια όσον αφορά την ε, διοικητική ικανότητα και όσον αφορά και τα προβλήματα των συνδικάτων ε, και των ενώσεων των εργαζομένων θα πρέπει επ' αυτόν ε, να εξετάσουμε να δούμε αν πρόκειται για θέματα συνδικάτων και που αφορούν και δικαιώματα εργαζομένων. Φυσικά πρέπει η νομοθεσία να ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς προδιαγραφές ε, για να διασφαλίζονται αυτές οι πτυχές. Τώρα, από πλευρά συναδέλφου, πάλι έγινε παρέμβαση για το διοικητικό από πλευρά ε, διακυβέρνηση ε, δυναμικό για μια μικρή τέτοια χώρα. Πρέπει είναι, να είναι σημαντικό. Δεν χρειάζεται να επινοηθεί, να επανεφευρεθεί ο τροχό. Πρέπει και σε σχέση και με την Κροατία να καταλήξουμε σε μια διευθέτηση αυτών των θεμάτων ώστε οι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων να καταλήξουν σε μια τέτοια τροχιά προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι αναφέρθηκε, αλλά για το κεφάλαιο 8, όταν έρθει η ώρα για Διαπραγματεύσει. θα είναι ένα ζήτημα για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις δεδομένων των ενισχύσεων στον τομέα του αλουμινίου έχει κλείσει, έχει πρόβλημα η βιομηχανική αυτή μονάδα, αναζητείται αγοραστής και πρέπει να δούμε και το πρόβλημα αυτό, διότι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης είναι προτεραιότητα οπωσδήποτε. Αναφέρθηκε το υψηλό ποσοστό ανεργίας. Έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα αυτό το σημείο. Εξαρτώνται από τον τομέα παροχής υπηρεσιών και τον τουρισμό φυσικά και η δημιουργία κάποιων θέσεων απασχόλησης στη βιομηχανία θα ήταν πολύ χρήσιμη υπόθεση. Τώρα, επίλυση μεθοριακών θεμάτων. Όταν πήγα εκεί το έθιξα σε ανώτατο επίπεδο με εκπροσώπους ε, κυβερνητικών κύκλων. Τώρα, για τις άδειε ε, αναζήτησης ε, πετρελαίου στις παράκτιες περιοχές στην Αδριατική θα πρέπει να δούμε εδώ μέσα σε ποιο πλαίσιο μπορούν να γίνουν όλα αυτά για την αναζήτηση πετρελαϊκών αποθεμάτων. Πρέπει όλα αυτά να διευθετηθούν με τον καλύτερο τρόπο ταχύτερα. Τώρα, σε σχέση με ε, την προσφυγή στο ε, Διεθνές Δικαστήριο, ίσως ε, μια διμερής επίλυση προβλημάτων μπορεί να ήταν πολύ χρήσιμη όσον αφορά εθνικούς ε, πόρους, ενεργειακούς πόρους και αποθέματα. Τώρα, μπορεί κανείς και οριζόντια, διασυνοριακά να κάνει κανείς εξόριξη αυτών των ενεργειακών αγαθών και αυτό περιπλέκει περαιτέρω τα θέματα. Από πλευρά συναδέλφου για την καταχώρηση ψηφοφόρων σε μητρώα και καταλόγους είναι πολύ σημαντικό για τις προεδρικές εκλογές που θεωρήθηκαν δίκαιες και δημοκρατικές. Όμως η καταχώρηση ψηφοφόρων πρέπει να γίνεται με δίκαιο και ορθό δημοκρατικό τρόπο. Οποιεσδήποτε προτάσεις σας θα εξεταστούν με ενδιαφέρον από μένα. Αναφέρθηκε και το θέμα της προστασίας ε, ατόμων και αυτό θα ληφθεί υπόψη. Κύριε Βουλιάνοβιτς, σας ευχαριστούμε για τα σχόλια κατά πολέμηση οργανωμένου εγκλήματος ε, και διαφθοράς. Για τον συνάδελφο Κούκαν, όλα τα σχόλια που έκανε τα δέχομαι και συμφωνώ με αυτά. Είναι πολύ σημαντικά μια, αυτά τα θέματα για μια μικρή χώρα όπω ε, το Μαυροβούνιο και που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει κάθε δυνατότητα δυνατότητα ε, από πλευράς ε, ε, ξένου συναλλάγματος. Καλωσορίζω τα θέματα τα οποία αναφέρατε εσείς συνάδελφε, δεν το είχα συνειδητοποιήσει αυτό και πολύ καλό αυτό. Κύριε Πίκουλα, αν... το θέμα είναι ότι εγώ πιστεύω ότι ήταν 5,5% Είδαμε σε σχέση με το, δημοψήφισμα για τη συνθήκη της Νίκαιας ένα τέτοιο ποσοστό διαφορά σε ένα δημοψήφισμα είναι μικρό αλλά παρόλα αυτά στέφθηκε με επιτυχία το δημοψήφισμα εκεί. Αυτά είναι τα ουσιοθέστερα στοιχεία. Θα τα συζητήσουμε όταν θα έχουμε τις τροπολογίες και θα δούμε και τις συμβαστικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ για τις προτάσεις σας συνάδελφοι. Σας ευχαριστούμε κύριε Τάνοκα. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για την έκθεση 5η Δεκεμβρίου 12 το μεσημέρι. Και ολοκληρώνεται αυτό το σημείο τώρα και περνάμε άμεσα στην έκθεση ή την ενημέρωση από την κυρία Γέγλε όσον αφορά την αποστολή στο Τατζικιστάν 7 ε, Νοεμβρίου 2013. Έχετε τον λόγο κυρία Γέγλε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Δεν είπατε πόσο χρόνο, πόσα λεπτά ή δευτερόλεπτα έχω στη διάθεσή μου πρόεδρε. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Ναι, χωρί όριο, αλλά εντάξει, λέει η κυρία Γέγλε, θα επικεντρωθώ και θα είμαι σύντομη στην παρουσίασή μου. Και θα παρακαλούσα και οι συνάδελφοι να παραμείνουν στην αίθουσα, γιατί έχουμε σημαντικά θέματα και να μην αποχωρήσουν. Το 2010 είχα πάει στο Τατζικιστάν για ε, επιτήρηση εκλογών με την αντιπροσωπεία μας. Από την 4η 7η Νοεμβρίου εφέτος ξαναπήγαμε εκεί διεξήχθησαν προεδρικές εκλογές. Οι συνάδελφοι ήταν από το ΕΛΚ, ο κ. Κασίνη από την Ιταλία, από τους σοσιαλιστές, η κυρία Τερέσα Αριέρα Μαδουρέλια από την Ισπανία, ο κ. Περόνι από την Ιταλία και ο συνάδελφος Γιώαχιμ Τσέλερ. Είχαμε ενταχθεί λοιπόν στον ΟΑΣΕ και στις ε, σχετικές αυτές ε, διακριβώσεις και δραστηριότητες και μπορώ με κάθε σαφήνεια να τοποθετηθώ και να πω ότι είχαμε καλή συνεργασία και συμβίωση μεταξύ μας. Όσον αφορά την επιτήρηση εκλογών δεν είναι πάντα αυτό δεδομένο και δεν είναι απλή υπόθεση. Είχαμε όμως ε, πολύ καλή επαφή και καλές σχέσεις και στο τέλος ε, οι αναλύσεις από πλευρά μας συνέπιπταν ε, επί των συμπερασμάτων μας. Ούτε σε ένα σημείο δεν παρεκκλίναμε ο ένας από τον άλλον. Φυσικά οι αρχές ε, ε, του ΑΣΕ για τις ε, δημοκρατικές εκλογές είναι δεδομένες. Υπάρχει δέσμευση για αυτές, τον σεβασμό αυτών των αρχών. Και αυτό οδηγεί να υπάρχουν κάποιες επικρίσεις για το ένα ή άλλο σημείο και που πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα για να βελτιωθούν και ελπίζουμε ότι θα βελτιωθούν όπως πρέπει. Επιπλέον τονίσαμε και κάτι ιδιαίτερα. Ήταν πολύ σημαντικό για την ενημέρωση αυτό. Είχαμε καλές συναντήσεις προς ενημέρωση και επικαιροποίηση με τις αρχές αρμόδιες ε, για την διεξαγωγή των εκλογών και με τα αντιπολιτευτικά κόμματα, με τις δύο κυριότερες ομάδες που στο τέλος τέλος ε, με <clears throat> την απαγόρευση συμμετοχής της υποψηφίου Social Democratic, Party, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και το κόμμα της Ισλαμικής Αναγέννησης αυτό οδήγησε σε επικρίσεις για το ότι δεν κατέστη αυτό εφικτό. Και σε συζητήσεις με τα άτομα αυτά, τους δύο προέδρους και την γυναίκα υποψήφιο που δεν επετράπει να συμμετάσχει στις εκλογές, κατέστη σαφές ότι χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι ότου να οριμάσουν τα πράγματα στο Τατζικιστάν και να μπορέσουν να λειτουργήσουν τέτοιες πρωτοβουλίες, ώστε τέτοιες ενώσεις, σύλλογοι και ομάδες εκπροσώπησης να μπορούν να εκπροσωπούνται και να μπορούν να κερδίσουν, να συνεισφέρουν σε μια πολιτική αντιπαράθεση που δεν μπορεί σήμερα πλήρως να διεξαχθεί και να διαμορφωθεί. Η υποψήφια απέναντί μου με κάθε σαφήνεια μου είπε είναι μια πολύ αξιόλογη και σεβάσμια καθηγήτρια στην πόλη του Σανμπέ. Είπε όμως ότι από πλευρά του Ισλαμικού κόμματος στην Ήπεθρο επειδή δεν φοράει μαντίλα δεν γίνεται αποδεκτή ως άτομο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθεί. Θέλω ρητά να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τους δικούς μας συνεργάτες που από το Κοινοβούλιο μας συνόδευσαν σε αυτό το έργο. Ήταν πάρα πολύ επικοδομητική η παρουσία τους και η συνεισφορά τους. Ήταν πολύ επικοδομητική η συνεργασία. Εμείς οι Ευρωβουλευτές μπορούσαμε πάντα να βασιζόμαστε το ότι τα πράγματα λειτουργούσαν καλά και πήγαιναν καλά χωρίς τριβές και προβλήματα. Και Περαιτέρω μεγάλες ευχαριστίες απευθύνω στην, προς την Ευρωπαϊκή ε, ε, το γραφείο που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση επιτόπου εκεί. Συνεισέφεραν πολλές πληροφορίες ε, να εισρεύσουν και να είμαστε εμείς αποδέκτες αυτών των πληροφοριών και τα πράγματα πήγαν καλά. Ο πρόεδρος Ραχμών με 83% των ψήφων επανεξελέγει. 83% ήταν κάπως μικρότερο αυτό το αποτέλεσμα σε ψήφους από ό,τι την τελευταία φορά. Αυτό που ήταν αξιοπρόσεκτο, αξιοπρόσεκτο είναι ότι Στι ε, τελευταίες, στις τελευταίες εκλογές ε, δεν ε, είχαμε ας το πω έτσι παρατυπίες ή δεν είχαμε κάποιους, ας κάποιες αμφισημίες. Μπορούσαν να τολμήσουν να πάνε εκλογής στα εκλογικά τμήματα και να διαγράψουν ένα, το όνομα ενός υποψηφίου ή να τοποθετηθούν υπέρ ενός άλλου χωρίς να φοβούνται. Και αυτό σε σχέση με τους συναδέλφους πρέπει να το αναφέρουμε όταν είναι κάποιοι μορφωμένοι άνθρωποι που ήταν υπεύθυνοι για την εκλογική διεργασία, ήταν πολύ σαφές ότι τήρησαν, τηρούσαν τις προδιαγραφές και ε, τις διατάξεις. Όσο περισσότερο όμως εκινείται κανείς στον χώρο της υπαίθρου, τόσο περισσότερες, ε, ας το πω έτσι, παρατυπίες σημειωνόντουσαν. Δηλαδή, θα ψηφίσω εγώ για όλη μου την οικογένεια. Εντάξει, τέτοιου είδου α το πω τοποθετήσει. Ε, ε, Κάποιο ε, αναλάμβανε τέτοιου είδου πρωτοβουλίε πηγαίνοντα στον εκλογικό θάλαμο για να ψηφίσει. Ήταν πολύ μικρά αυτά τα, αυτές οι καμπίνες. Με πέντε διαβατήρια ήρθε κάποιος πέντε ταυτότητες. Έπρεπε και για τη γυναίκα του και τις κόρες του να ψηφίσει και είπε «Ε, αυτές έπρεπε να εργαστούν και ήταν απασχολημένες, έρχομαι εγώ να ψηφίσω για λογαριασμό τους. Ίσως αυτό θα πρέπει να το δούμε σε μια πιο μακροχρόνια προοπτική για να αλλάξουν κάποια πράγματα στο Τατζικιστάν. Είχαμε και μια κοινή δήλωση προς τον τύπο και θέλω να το τονίσω αυτό από πλευράς ΟΑΣΕ και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κρούσαμε κόδωνα κινδύνου και τονίσαμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Απαιτήσαμε να διεξαχθεί μια πολιτική συζήτηση που θα πρέπει να διεξαχθεί σε αυτή τη χώρα. Οι νέοι άνθρωποι να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδου διαβουλεύσεις και συζητήσεις. Κάτι τέτοιο δεν πρέπει πια να είναι δύσκολο Θέλουν οι νέοι να γίνει αυτό. Και αυτό είναι το ζήτημα. Πρέπει να γίνει αυτό. Και είπαμε προς την αντιπροσωπεία μας να κάνουμε πάντα τέτοιες προτάσεις ώστε να προαχθούν αυτά τα θέματα. Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες. Να μην δίνεται εξουσιοδότηση σε κάποιους να πηγαίνουν να ψηφίζουν εξ ονόματός τους. Να συμμετέχουν οι ίδιες στις διαδικασίες. Και ολοκληρώνω τώρα. Από το 2010 άλλαξαν κάποια πράγματα άλλαξαν. Μάλιστα. Δεν άλλαξαν επαρκώς και δεν ήταν επαρκείς οι μεταβολές και οι αλλαγές. Πρέπει όμως να το δούμε ότι οι άνθρωποι που έχουν 1300 χιλιόμετρα σύνορα προς το Αφγανιστάν ζουν σε σύνορα τα οποία δεν είναι ασφαλή, απόλυτα ασφαλή, δεν μπορούν να εποπτεύονται με, ε, με τον ασφαλέστερο τρόπο. Υπάρχουν φοβίες ε, και φόβοι Βασίζονται στον ε, Ραχμόν οι πολίτες του Τατζικιστάν για όσα έκανε και την προσπάθεια που ανέλαβε να υπάρξει μια ε, κοινή ανάπτυξη των εντελώς διαφορετικών εθνοτικών ομάδων. Και αυτό ικανοποιεί αυτέ τι ομάδε και του το αναγνωρίζουν με ιδιαίτερο τρόπο και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό, αφού αυτή είναι η θέση, η θέση τους. Θα ήθελα σε τέτοιου είδου επιτηρήσει εκλογών να δραστηριοποιούμαστε ενεργά. Εκεί μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει το πρόσωπό τη την ταυτότητά τη ευδιάκριτα για τι αρχέ και αξίε μα. Μπορούμε να καταβάλουμε προσπάθειες ενεργά. Έτσι λοιπόν οι αντιπροσωπείε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητε να μα εκπροσωπούν σε αυτέ τι χώρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρο σα ευχαριστώ θερμά κυρία Γέγκλε. Και από πλευράς μου ίσως μια πολύ σύντομη ερώτηση. Πώς έχουν οι σχέσεις με τη Ρωσία σε σχέση με το Τατζικιστάν και την ιδέα από τη Ρωσία για μια τελωνιακή ένωση που εκινεί από την Μόσχα και που προωθεί η Μόσχα ιδιαίτερα ενεργά. Τι γίνεται στο Τατζικιστάν. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις ή συζητήσεις ως προς αυτό το θέμα, προς αυτή την κατεύθυνση. Η κυρία Γέγλε. Είμαι μέλος της αντιπροσωπείας για τις χώρες της Κεντρικής Ασίας από τη δεκαετία του 90. Γνωρίζω τις χώρες αυτές πολύ καλά. Το σύνολο των, των περιφερειακών αυτών χωρών και το Τατζικιστάν βασίζονται και θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι εταίρος τους στη μέση ενδιάμεσα μεταξύ Κίνας που κάνει πάμπολες προσπάθειες, διαθέτει δυνατότητες κονδύλια και της Ρωσίας ε, και τον είπα από την άλλη πλευρά. Αλλά της Ρωσίας κυρίως από την άλλη πλευρά. Αναμένουν από εμάς ένα διαμεσολαβητικό ρόλο. Όχι υποχρεωτικά περισσότερα κονδύλια από εμάς. Αναμένουν όμως μια εσωτερική, ψυχολογική θα έλεγα υποστήριξη που μπορούμε σίγουρα να δώσουμε και δίνουμε. Το πρόβλημα όμως στην περιφέρεια αυτή ποιο είναι οι πρόεδροι ε, Ναζαρμπάιεφ, Καριμόφα ε, ε, δεν μπορούν να συζητήσουν ένας με τον άλλον. Κάνουν λόγο ο ένας για τον άλλον, αλλά δεν συζητούν μεταξύ τους. Ακόμα και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Είναι πρόβλημα το ότι δεν συζητούν ανοιχτά μεταξύ τους. Έχουμε εδώ έργο που πρέπει να επιτελέσουμε για το σύνολο των χωρών της Κεντρικής Ασίας, για όλες τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες και χώρες. Έχουμε ιδιαίτερες ευθύνες και ρόλο για το Τατζικιστάν που έχει αυτά τα μακρά σύνορα με το Αφγανιστάν. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε περισσότερα, να, περισσότερο, να κάνουμε περισσότερα πράγματα εκεί. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν από δύο χρόνια Είχαμε ένα φράγμα το οποίο μας πήγαν να δούμε γιατί ήταν ενδιαφέρον και ήθελα να το δω. Από τον Τουσανμπέ πάει κανείς μέσω ε, ενός διάσελου σε μια ε, ε, κοιλάδα και φοβόμαστε ότι δεν θα καταφέρναμε σε μια μέρα με τέτοιες αποστάσεις. Ξαφνικά, να και μια σύραγγα, ωραία, και οδικά μπορούσε κανείς να διαβεί από εκεί. Μου είπαν η Κίνα μας τα πλήρωσε αυτά και μας έδωσε τα κονδύλια να γίνουν αυτά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κάποιες άλλες προδιαγραφές και απαιτήσει. Δηλαδή εμείς δεν ήταν δυνατό να πληρώσουμε αυτή τη σύραγγα, ούτε μπορούμε ούτε ήταν δυνατό να την πληρώσουμε. Έχουμε τεράστιο έργο να επιτελέσουμε. Αλλά να αναζητήσουμε επαφές, να γίνει κατανοητό ποιε είναι οι θέσεις μας. Γιατί θέλουμε να ειρηνεύσουν, να οδηγηθούν σε ειρήνευση οι χώρες αυτής της περιφέρειας, αυτής της περιοχής. περιοχής. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνίστρια, ανταγωνιστικοί δύναμη έναντι της Ρωσίας. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να είμαστε όμως εταίροι για αυτές τις χώρες. Αυτό αναμένουν από εμάς εκεί επιτόπου οι πολίτες. Πρόεδρο σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γέγλερ. Και έτσι ολοκληρώνουμε τώρα και αυτό το σημείο. Και έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε και να, με την ημερήσια διάταξη και τα θέματά μας. Το επόμενο σημείο τώρα είναι η ανανέωση <clears throat> της Συμφωνίας Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας για θέματα επιστήμης και τεχνολογίας. Εισηγητής ο κύριος Ρούτσεκ. Θα ήθελα τώρα να του δώσω τον λόγο του κύριου Ρούτσεκ. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. It's... Πρόεδρε, είναι η γνωμοδότησή μας για την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορία. Αφορά ακριβώς την ανανέωση της Συμφωνίας Συνεργασίας στην επιστήμη και στην τεχνολογία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η συμφωνία συνήφθη το 2000, ανανεώθηκε για 5 έτη το 2009, συνεπώς η πρόταση αφορά την περαιτέρω ανανέωση για επιπλέον 5 έτη στην παρουσία της μορφή. Ο στόχος είναι να εντείνουμε περαιτέρω τις διεθνείς, τις διμερείς με σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η εμπειρία είναι θετική ως τώρα, παρά τις πολλές δυσκολίες που είχαμε με την Ρωσική Ομοσπονδία. Μάλιστα τις τελευταίες μέρες είχαμε το θέμα της Ουκρανίας και την πίεση της Ρωσίας στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Παρά τα προβλήματα αυτά λοιπόν, σε πολλούς τομείς επιστήμης και τεχνολογίας μπορούμε να συνεργαστούμε ικανοποιητικά προς αμοιβαίο όφελος στον τομέα της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. Για όλους αυτούς τους λόγους, καλό την ε, Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή να εγκρίνει την ανανέωση αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Ρούτσεκ, θέλει κανείς το λόγο. Οπότε, η ψηφορία θα γίνει 12 Δεκεμβρίου στην Αρμόδια Επιτροπή, στην Ήτρε 17 Νοεμβρίου στην Επιτροπή Τεχνολογίας και Ερευνές. Οπότε κλείσαμε με την ημερήσια διάταξη. Ανακοινώνω ότι το επόμενο ζήτημα στη ημερήσια διάταξη ενημέρωση από τον αντιπρόεδρο της αντιπροσωπείας για την Μιανμάρ αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση μας στο Στρασβούργο. Οπότε θα τα ξαναπούμε σήμερα το απόγευμα στις 3. Ε, Καλό μεσημέρι.